Der Präsident! Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Ε, αρχίζει πάλι η συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε. Τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Ισοβίου Γερουσιαστή καθηγητή Μόντι, Πρόεδρου του Συμβουλίου της, των Υπουργών της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Μόντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τιμή που σας έχουμε μαζί μας και σας καλωσορίζω θερμά εξ ονόματος ολόκληρου του σώματος. Κυρίες και κύριοι, Δύο λόγια διαδικαστικά. και ήθελα να πω στα μέλη ότι δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye εδώ, οπότε δεν έχει νόημα να ανέβετε με τα λευκά φύλλα, δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye. Το λέω αυτό γιατί ε, έχω πίσω μου πολλές διαδικασίες Catch the President. Ε, πολλοί ήθελα να μου συστήσουν το Catch the Eye και για αυτή τη διαδικασία, αλλά δυστυχώς δεν προβλέπεται τελικά. Θα ήθελα να μιλήσω να ε, δώσω το λόγο για το θέμα αυτό της οικονομικής κρίσης ανάπτυξης και απασχόλησης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Μάριο Μόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και για την Ιταλική κυβέρνηση το ότι με προσκαλέσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά σας για να εκφράσω και να πω μερικά λόγια. Καταρχήν θα ήθελα να τιμήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα αποτελεί μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντήθηκα με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 1995 για τις ακροάσεις στα πλαίσια των ακροάσεων για τους επιτρόπους για δέκα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν για μένα βασικός και αποφασιστική σημασία συνομιλητής και ήταν να εξελίσσεται η δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και να ε, επαυξάνεται και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να χαιρετήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο βασικός φορέας για να αναπτυχθεί ο εκδημοκρατισμός και η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βρίσκομαι σε ένα διαφορετικό έδρανο, εδώ ενώπιόν σας και μπορώ να σας πω ότι είναι αλληλένδετες αυτές οι ευθύνες. Νιώθω μεγάλη ευθύνη έναντι της χώρας μου και έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλές φορές είδα από τις Βρυξέλλες ως επίτροπος εθνικές κυβερνήσεις που έδρασαν ως κατήγοροι των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης αφού συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων στα θεσμικά αυτά όργανα. Εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου ποτέ να μην παίξω αυτό το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. E Και εξηγώ στους συμπολίτε μου πάντα ότι έχουν γίνει μεγάλες θυσίες. Έχουμε να κάνουμε με δύσκολες μεταρρυθμίσεις, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν οι Ιταλοί σήμερα. Δεν επιβάλλονται όμως από την Ευρώπη. Είναι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και για την κοινωνία των πολιτών και έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά μας. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τις αποφάσεις τις λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ καθοδηγώ μία χώρα, βρίσκομαι στο πιδάλιο μίας χώρας, όπου υπάρχει μια κοινή γνώμη υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οικοδόμησης. Πρόκειται για κάτι σπάνιο. Αυτή λοιπόν την πρώτη ύλη θα την καλλιεργήσω περαιτέρω και νομίζω ότι θα πρέπει με μεγάλη φροντίδα να πείσω τους συμπολίτε μου με ακλόνητα επιχειρήματα. Και σε κάθε ευκαιρία καλό και άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν την ίδια επιρροή ως προς το κοινωνικό αυτό οικοδόμημα. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, δίνει μεγάλο αγώνα για να βγει από την κατάσταση επίγουσας ανάγκης. Νομίζω ότι βαθμία το κατορθώνουμε. Η χώρα μας θα βγει από αυτή τη μεγάλη σκιά στην οποία βρισκόταν και δεν θα αποτελέσει αιστεία μετάδοσης αυτού του κινδύνου στην Ευρωζώνη. Καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής παγιοποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το καλοκαίρι, ο προκάτοχός μου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ανέλαβε την ευθύνη να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά μας και το 2013 να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας δύο χρόνια πριν από την υποχρέωση, την κοινοτική μας. Η κυβέρνησή μου επανέλαβε αυτή τη δέσμευση. Δεν ζήτησε εξαιρέσεις, αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να προσδώσουμε το 5% του ΑΕΠ για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να, φτάνουμε, να φτάσουμε στους στόχους, δηλαδή να ανταποκριθούμε στα δημοσιονομικά, στις δημοσιονομικές απαιτήσεις. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχει ένας συγκερασμός δυνάμεων έτσι ώστε να φτάσουμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν πρόκριμα για να βγούμε από την κρίση. Βρισκόμαστε σε μία οδό ασφάλειας και εξασφάλισης. Υπάρχουν πολλά ενθαρρυντικά στοιχεία και δεν θα περιοριστούμε να δεχτούμε παθητικά τις πολιτικές κατευθυντηρίες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμές και να διαδραματίζουμε το ρόλο που αρμόζει σε μία από τις μεγάλες ιδρύτριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ε, in questo... Υπ' αυτή την έννοια, με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση αυτή για στενή συνεργασία που προήλθε από την Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο και σε αυτή την τριγωνική σχέση είπα ότι η Ιταλία θα συνεισφέρει για την ανέλυξη της ε, κοινοτικής μεθόδου γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να δημιουργήσουμε γέφυρες και όχι προσκόμματα και στεγανά για τις χώρες που δεν βρίσκονται ακόμα στην Ευρωζώνη. και που κάποια στιγμή θέλουν να προσχωρήσουν. Δεν είναι από τις χώρες που δεν το επιθυμούν. Θα πρέπει η Ευρώπη να μην αποκλείει, αλλά να συνενώνει. Επειδή μας απασχολεί η οικονομική κρίση, η ανάπτυξη και η απασχόληση, θα ήθελα να μιλήσω για τους βασικούς κινδύνους αυτής της φάσης που διανύουμε το ευρώ αποτέλεσε το πιο φιλόδοξο και το πιο τελειοποιημένο στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής ζωής. Δεν θα πρέπει όμως να αποτελέσει στοιχείο αποδυνάμωσης και διχασμού της Ευρώπης, καθώς και κατακαιρματισμού, κατακαιρματισμού της. Ελπίζω και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επιληθεί η κρίση στην Ευρωζώνη, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε εξίσου προσπάθειες για την ανάκτηση ενός ε, ενωτικού πνεύματος. Η κρίση της ε, Ευρωζώνης οδήγησε σε πολλές ε, μνησικακίες και στερεότυπα δίχασε τους Ευρωπαίους ανάλογα με το γεωγραφικό τους ε, μήκος και πλάτος σε περιφερειακά κράτη και κράτη του κέντρου. Αυτές οι υπεραπλουστεύσεις θα πρέπει να εξαλειφθούν. Εκπρόσωπο μία χώρα που θεωρείται περιφερειακή από γεωγραφικής πλευράς και δεν με ενοχλεί αυτή η θεώρηση πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι κράτος του κέντρου ήταν και η Ιταλία από πλευράς ε, λήψεως αποφάσεων. Αλλά τα κράτη του κέντρου, η Γερμανία και η Γαλλία, ε, αποτέλεσαν, βρίσκονταν και στο κέντρο της ε, κρίσης ως προς το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2003, όταν υπό Ιταλική Προεδρία, μάλλον ε, Ιταλική Προεδρία και στο ΕΚΟΦΗΝ, οι δύο αυτές χώρες άσκησαν την πολιτική τους επιρροή σε άλλα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην ισχύσει ο μηχανισμός ε, σταθερότητας. Αυτό το αναγνωρίζουν σήμερα και η Γαλλία και η Γερμανία. Δεν ε, λέω λοιπόν τίποτα το μη γνωστό ή και το όχι τόσο ευχάριστο προς την καγκελάριο και τον πρόεδρο της Γαλλίας. Αλλά αυτό το βούλνους προήλθε από εκεί. διότι μιλούσαμε για μία δημοσιονομική πειθαρχία που στη συνέχεια δεν τηρήθηκε. Άρα και το κέντρο φέρει ευθύνες όπως και η περιφέρεια. Και πολλά κράτη της περιφέρειας ε, φέρουν ευθύνη όπως το κράτος το οποίο τώρα εκπροσωπώ. Γιατί αντί για πειθαρχημένοι ήμασταν απίθαρχοι ως προς τα δημοσιονομικά μας. Δεν πρέπει όμως να μιλάμε για καλούς και κακούς. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και για το παρελθόν και για το παρόν. Ε, Χρειάστηκαν οκτώ επίπονα χρόνια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή Καταρχήν η Επιτροπή, και αυτό το υπογραμμίζω, γιατί πρόκειται για την οστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα θεσμικά όργανα, λοιπόν, για να επανέλθω, για οκτώ χρόνια ασχολήθηκαν για να επανικοδομήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χρειάστηκαν οκτώ επίπονα χρόνια γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση των έξι νομοθετημάτων του Six που έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία από εκείνη του Συμβουλίου. Άρα στην ιστορική αυτή φάση, εάν μιλάμε για απειθαρχία ως προς το εκτελεστικό σκέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο απετέλεσε παράγοντα πειθαρχία εξαιτία και χάρη μάλλον στην προσπάθεια που κατέβαλε, στην επίπονη προσπάθεια που κατέβαλε. νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αποδώσουμε ευθύνες και να μιλήσουμε για το πέρασμα σε μία άλλη σελίδα ανάπτυξης. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε και τα δύο σκέλη και στην καθημερινή μας ζωή το βλέπουμε αυτό. Χτες χρειάστηκε να λάβουμε μία δύσκολη απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών της Ιταλίας. Δηλαδή, δεν μπορέσαμε να δεχτούμε να είμαστε υποψήφια χώρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη. Υπήρξε μεγάλη απογοήτευση από την Ρώμη ιδιαίτερα και από τους Ιταλούς γενικότερα, αλλά νομίζω ότι η κοινή γνώμη της Ιταλίας καταλαβαίνει πολύ καλά ότι υπάρχουν άλλες επιτακτικές ανάγκες. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον μου δόθηκε για άλλη μια φορά το στίγμα ότι η Ευρωζώνη είναι ύψης της σημασίας για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Αφήνουμε λοιπόν για αφήνουμε παρόμοια θέματα για το μέλλον και αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι δεν μπορούμε να μεταθέτουμε ευθύνες για το μέλλον και για τις μελλοντικές γενές. Η Ιταλία συνεισέφερε στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε ευρωπαϊκούς αγώνες και εκδηλώσεις, αλλά νομίζω ότι τέτοιες μαρτυρίες είναι σκόπιμες για, τα, να κατανοήσουμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ύψης της σημασίας και προέχει όλων, όλων των άλλων δραστηριοτήτων επιτάπητος, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μιλάμε για ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο στο μέλημα της Ιταλίας, γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την δημοσιονομική μας πειθαρχία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου και στη συνέχεια της 1ης Μαρτίου θα ασχοληθεί με θέματα ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να περάσει στην καθημερινή μας εργασία. Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρόκριμα της ανάπτυξης. Η Ιταλία ζήτησε και έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία υψηλότερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη μεταξύ των οικονομικών στόχων. Αυτό είναι δυνατόν χωρίς να αμφισβητηθεί η πειθαρχία και αρκεί να βγούμε από ορισμένους κοινούς τόπους. Δηλαδή, η ενιαία αγορά έχει πολλά να πει και να κάνει. Ο Επίτροπος Μπάρνιε ηγήθηκε της τελευταίας προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή της πράξης για την ενιαία αγορά. Και εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα για να ανταποκριθούμε και έμπρακτα σε αυτό μέσα στα πλαίσια του ορίζοντά μας έτσι ώστε η ενιαία αγορά να μην είναι ένα συμπίλημα οδηγιών και κανονισμών. Αποτελεί το κόρπους και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να προωθηθεί. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είχα τονίσει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δημοσιονομικά μας, τη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά δεν θα πρέπει να γίνει το ίδιο και για την Οικονομική Ένωση, για την ενιαία οικονομική αγορά. Γιατί θα πρέπει να μιλάμε για μηχανισμούς με κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κράτος μέλος το οποίο παραβιάζει τους κανόνες, να τους παραβιάζει για τέσσερα με πέντε χρόνια έως ότου προσφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία δυσλειτουργίας και των οικονομικών και της Ευρωζώνης. Έχουμε προσδώσει μεγάλη σημασία στην Νομισματική Ένωση, όμως δεν προσδώσαμε την ίδια σημασία στην Οικονομική Ένωση, που είναι το υπόβαθρο της Νομισματικής Ένωσης. Θα πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία και σε αυτό το σκέλος, το καθαρά οικονομικό. Δεν θα μακρηγορήσω θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ πειθαρχημένο ως όπως είσαστε και εσείς στην κατανομή του χρόνου. Θα ήθελα να μιλήσω για τα stability bonds, για τα ομόλογα σταθερότητας. Αποφανθήκατε θετικά με μεγάλη πλειοψηφία και εγώ έχω προωθήσει αυτή την έννοια. Δεν θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα στοιχεία απειθαρχίας, αλλά πειθαρχίας και ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών. Με βάση την πράσινη βίβλο της Επιτροπής και το ψήφισμά σας που εγκρίνατε σήμερα, έτσι ώστε να είναι πιο πειθαρχημένες οι χρηματοπιστωτικές αγορές έναντι των κρατικών προϋπολογισμών. Είναι ένα από τα μέσα τα οποία θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη και ιδιαιτερότητες. Εάν μια χώρα θεωρεί ότι τα ομόλογα σταθερότητας θα πρέπει να προτρέξουν των αναγκών, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθει η χρονική στιγμή όπου θα τα επανεξετάσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για τις οικονομικές επενδύσεις και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για την έννοια του fiscal compact και μιλάμε για ισοσκελισμό των προϋπολογισμών μας. Θα έπρεπε να μιλούσαμε περισσότερο για χρυσό κανόνα, για golden rule. Αλλά και στη γερμανική οικονομία, όπως ξέρετε, ο χρυσός κανόνας, το golden rule, όριζε τα πάντα. Δηλαδή, μιλούσαμε για κρατικό χρέος, αλλά μιλούσαμε κυρίως για επενδύσεις, για επενδύσεις στα πλαίσια της κεφαλαίου αγοράς. Κάποια μέρα η Ευρώπη αφού θα μετασχηματιστεί κάτι το οποίο καταφέραμε με βάση την κουλτούρα της Γερμανίας, κάποια μέρα θα μπορέσουμε να προβάλλουμε και άλλα αναπτυξιακά μέσα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άρθρο που είδα στο γερμανικό, γαλλικό και ιταλικό τύπο που προσυπογράφω και εγώ μαζί με την ε, Σιλβί Γκουλάρ. Χρειαζόμαστε και ανάπτυξη αλλά και δημοκρατία, από την οποία δεν μπορούμε να παρετηθούμε. Πώς μπορούμε να συσχετίσουμε δημοκρατία και ολοκλήρωση. Νομίζω ότι συμφιλιώνονται η ολοκλήρωση, η οικονομική ολοκλήρωση και η δημοκρατία. Συνεχίζει ο Πρωθυπουργός Μόντι στα Ιταλικά, στα Αγγλικά διότι ε, μόνο μία επιφανειακή νησιωτικού τύπου πολιτισμική θεώρηση θα μπορούσε να θεωρήσει να θα μπορούσε να θεωρούσε ότι η ολοκλήρωση σημαίνει υπερκράτος. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με παθιάζει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν σημαίνει υπερκράτος, super state. Μιλάμε και για την επικουρικότητα και για επικουρικότητα, η οποία όμως πρέπει να συμφιλειωθεί με τις αρχές της δημοκρατίας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται εις βάρος της δημοκρατίας. Δεν εφήβραμε τον τροχό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θεσμικό όργανο που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Εγώ συμμετείχα πολλές φορές στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το έδρανο της Επιτροπής. Ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάντα πολύ αυστηρός και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε άκρος αποτελεσματικοί υπό τη μεγάλη όθηση που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια μεγάλη εφεύρεση ενός μεγάλου πνεύματος του Ζαμονέ και πιστεύω ότι η έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημοκρατίας είναι δύο έννοιες πλήρως εναρμονισμένες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης της Ιταλίας. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε το άρθρο που δημοσιεύσατε μαζί με τη συνάδελφο Γκουλάρ Θα ήθελα για το άρθρο αυτό να σας ευχαριστήσω και τους δύο εξ ονόματος του σώματος. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη σύμπτωση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Και τώρα για πέντε λεπτά ο κύριος Ντόλα από το Λαϊκό Κόμμα. Κύριε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μόντι, συνάλφη. Ε, είμαστε πεπισμένοι όλοι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξηγιάνει τα οικονομικά της και να ξαναβρει το δρόμο της ανάπτυξης, αυτό που μας είπατε και εσείς πριν από λίγο. Θα ήθελα να σας πω αγαπητέ κύριε Μόντι ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες ξεκινήσατε εσείς στη χώρα σας δίνουν το παράδειγμα και στις δύο αυτές κατευθύνσεις αφενός ε, προεβείται σε μεταρρυθμίσεις σχετικά με θέματα τα οποία, ε, τα οποία δεν είχαν απασχολήσει προηγούμενες κυβερνήσεις και από την άλλη μεριά επιφέρατε σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Όλα αυτά δένουν προς την σωστή κατεύθυνση γιατί θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ε, και θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Χάρη στην εισαγωγή μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας θα γίνει αυτή η αγορά πιο δυναμική και ταυτόχρονα προστατεύει τους εργαζόμενους περισσότερο. Ε, καταπολεμάται επίσης τη διαφθορά, είστε υπέρ ενός πιο διαφανούς φορολογικού συστήματος και αυτά είναι σωστά γιατί θα ε, μειωθεί το φορολογικό βάρος που βαρύνει τους Ιταλούς. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό το πακέτο μέτρων που επαναλαμβάνω αποτελεί υπόδειγμα και παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Ελπίζω θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας και πολλές άλλες χώρες. Γιατί για να ξαναβρούμε την ανάπτυξη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα πολιτικό και οικονομικό κλίμα υπέρ της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε ελπίδα στους συμπολίτε μας, όχι μια ψεύτικη ελπίδα έτσι ώστε να απογοητευτούν γρήγορα. Θα πρέπει να είναι μια ελπίδα που θα βασίζεται στην ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένη σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα ευνοούν την κοινή μας ζωή. Η Ιταλική οικονομία είναι ισχυρή γιατί βασίζεται σε μια πραγματική οικονομία πάνω σε οικονομικούς τομείς και κλάδους ανταγωνιστικούς. Εσείς ε, πρέπει να βελτιστοποιήσετε αυτό το δυναμικό, να προχωρήσετε σε περαιτέρω φιλελευθερωποίηση οικονομίας και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι επίσης, να πάρουμε παράδειγμα από εσά. Θα πρέπει με τις εθνικές πολιτικές αλλά και τις ευρωπαϊκές πολιτικές να προωθήσουμε την χρήση των πόρων που υποχρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, τους ερευνητές και τα εκατομμύρια των νέων πολιτών που βρίσκονται σε ενεργεία να τους επιτρέψουμε να αναπτύξουν το δυναμικά τους. Αυτό ε, απαιτεί πνεύμα ευθύνης. Αυτό το πνεύμα το οποίο δείχνετε εσείς κύριε Μόντι αυτή τη στιγμή. Για ορισμένους ο πειρασμός είναι ψηλό ε, να συνδέσουν τα, τις δημόσιες δαπάνες και τις επενδύσεις. Όμως, χάρη στις επενδύσεις θα εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο προηγούμενος πρόεδρος της, ε, ε, ένας παλιότερος πρόεδρος τη Κομισιόν, ο κ. Δελόρ, είπε ότι δεν είμαστε ε, δεν ε, είμαστε ερωτευμένοι με την εσωτερική αγορά και ούτε με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα έλεγα εγώ στις 15 Φεβρουαρίου όμως οι προσπάθειές σας βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και μειώνουν την ανεργία. Ε, χρειάζεται να δώσουμε μια καινούρια ανάσα για την ε, ολοκλήρωση των ε, αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να μιλήσω επίσης ε, για την ενιαία εσωτερική αγορά η οποία 20 χρόνια μετά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ξέρετε όλοι πώς είμαι υπέρ της ατμομηχανής της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όμως θέλω και άλλες χώρες όπως η Ιταλία να ε, αυξήσουν το βάρος τους στην Ευρώπη. Επίσης θέλω να υποφελθώ τις ευκαιρίες για να χαιρετήσω την, ε, τη, τη στάση σας υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, γνωρίζετε ότι η επιστροφή στην διακυβερνητική μέθοδο θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Είναι σαν να επιστρέφουμε προ τα πίσω για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να χρησιμοποιήσετε το βάρο που έχετε έτσι ώστε να διαφωνήσετε και ε, με αυτή την ε, οπισθοδρόμηση. Το Κοινοβούλιο θα σας υποστηρίξει. Επίσης, το Κοινοβούλιο θέλει μια Ευρώπη αλληλέγγυα και υπεύθυνη. Μια Ευρώπη ολοκληρωμένη και μια πολιτική Ευρώπη. Νομίζω ότι με εσά ε, παρόντα βασιζόμαστε σε ένα σύμμαχό μας. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριο Σβόμποντα για έξι λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλώ ήρθατε στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο ε, εξ ε, των ε, Ιταλών Δημοκρατών, αλλά όλων των Σοσιαλδημοκρατών. Είπατε ότι εκλεγήκατε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ε, ε, μετά το λόγο σας που μόλις ακούσαμε θα σας εκλέγαμε ε, ευχαρίστως όλοι. Ε, γι' αυτό λοιπόν καλό είναι κάποια στιγμή να έρθετε και σε εμά. Οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλές και στην Ιταλία και στην Ευρώπη και ημών και της κοινή γνώμης. Μιλήσατε για την απασχόληση και το συνδυασμό της με δημοσιονομική πειθαρχία. Θα έλεγα κάνοντας ένα βήμα παραπέρα ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, αν υπάρχει ανάπτυξη και απασχόληση, επιτυγχάνεται ευκολότερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε ακούσει πολλές δηλώσεις και από την Ιταλία και από άλλες χώρες, αλλά ακόμη περιμένουμε την, τις πράξεις. Θέλω να παραθέσω ε, από την τελευταία σύνοδο κορυφής ε, και τον πρόεδρο Σαρκοζή που λέει ότι η απασχόληση πρέπει να είναι στην καρδιά όλων των πολιτικών μας ούτως ώστε να έχουμε μεγέθυνση, ανάπτυξη και ισορροπημένη, ε, ισόρροπη αηφόρο ε, ανάπτυξη λόγια που είναι οι πράξεις όμως μιλήσατε για τα ομόλογα σταθερότητας και άλλα μέσα. Συζητούμε για τις διάφορες πολιτικές για την ανάπτυξη, χωρίς δράση όμως. Δεύτερον, για μας ε, η κοινωνική Ευρώπη, ξέρετε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επίσης έχουμε την δήλωση του Συνόδου Κορυφής των, του G20. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη της κοινωνικής προστασίας σε κάθε χώρα μας. Είμαστε πεπισμένοι για τον ουσιαστικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα συζητήσαμε για τον κοινωνικό διάλογο και πώς, ε, για παράδειγμα, αποσαφρώνεται στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η Τρόικα λέει όχι κοινωνικός διάλογος, όχι κοινωνική εταίρη, μόνο νομοθετικά μέτρα και μετά κάποια στιγμή θα ε, ξανασυζητήσουμε για τη δημοκρατία. Για μας οι κοινωνικές πολιτικές και η ανάπτυξη μαζί με την δημοσιονομική πειθαρχία συμβαδίζουν. Δεύτερο θέμα για τους φόρους. Για την κοινωνική Ευρώπη το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να είναι κοινωνικό και δίκαιο και θα πρέπει να δώσουμε μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Και πάλι οι G20 λένε αναλάβουμε δέσμευση να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά μας ε, και τα ε, δημοσιονομικά συστήματα από τις παραβιάσεις ε, και τις λανθασμένες νομοθετικές δράσεις. Δεν λέει τίποτα για τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή. Τι θα πιστέψουν οι Έλληνες όταν τα χρήματα που πηγαίνουν στην Ελβετία δεν φορολογούνται ενώ εκείνοι θα πρέπει να μειώνουν φόρους για τα μειωμένα εισοδήματα, μισθούς και ε, εισοδήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για μα. Συχνά λέμε ότι ε, πρέπει να ε, δούμε τη φοροδιαφυγή. Η μελέτη από τις ομάδες μας δείχνει ότι αν εφαρμοστεί σωστά το, το φόρος αυτός, η φοροδιαφυγή δεν ε, ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Υπάρχει φοροδιαφυγή προς την Ελβετία, ε, και, τις Μπαχάμες και άλλες χώρες. Εκεί είμαστε... πιο ελαστικοί ενώ στα, στις χώρες μας όχι. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Η, η εξυγίανση σε μια ε, Ευρώπη με λιγότερη ανεργία, περισσότερε θέσει εργασία, με κοινωνικό σύστημα δίκαιο και φορολογικό σύστημα δίκαιο, μια τέτοια ε, δημοσιονομική εξυγίανση είναι ε, σωστή και θα γίνει δεχτή και από του πολίτε. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα οποία θα συμβάλλουν στη δική μα αντίληψη για την ανάπτυξη, όπω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα Επενδύσεων. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί να μην μην δώσει περισσότερα δάνεια σε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εκείνη μπορεί να δημιουργήσει ε, ανάπτυξη. Όσο για την Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος ε, Ντράγκη κάνει καλή δουλειά και ε, Θέλουμε ε, να συνεργαστούμε όλοι για να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα και δημιουργία ε, ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν με τους δύο Ιταλούς σε κεντρικές θέσεις, Μόντι, ε, Τράγκη, έχουμε ίσως μεγαλύτερες πιθανότητες για καλύτερες λύσεις. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Τελευταίο για τη Δημοκρατική Ευρώπη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η δημοκρατία και η ολοκλήρωση δεν αποτελούν αντίφαση. Η δημοκρασία για μας όμως δεν είναι το Συμβούλιο το ίδιο, γιατί κάποια μέλη του Συμβουλίου προσπαθούν να ανακτήσουν εξουσία, μεγαλύτερη δύναμη. Πολλοί πολίτες ε, λέγουν γιατί ε, ποιος θα είναι ο ρόλος ε, μετά την συνθήκη της Λισαβόνας του Κοινοβουλίου. Βεβαίως ε, μπορεί να μην ήταν προσφυλής συνθήκη για πολλούς κυβερνήσεις, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί το αίτημα του Κοινοβουλίου να είναι μέρος του, της δημοκρατικής αυτής διαδικασίας και όχι να ε, είναι παραγνωρισμένο. Μπορούμε να ε, επιφέρουμε αλλαγές αν συμμετέχουμε στις συζητήσεις από την αρχή. Επίσης δεν περιορίζεται η δημοκρατία στην Κομισιόν, ούτε ε, είναι σωστό εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων να παρεμβαίνουν σε επίπεδο κρατών μελών και να πολλές φορές αντί να βελτιώνουν να επιδεινώνουν την κατάσταση όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν υψηλές προσδοκίες από εσάς και σε σχέση με την δημοσιονομική σταθερότητα. Χαιρόμαστε που ήρθατε, δουλεύετε για μια ισχυρή Ιταλία και μια ισχυρή Ευρώπη. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε η Ιταλία ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ισχυρή, δημοκρατική, οικονομικά ασφαλής, ε, υγιής, με κοινωνική πολιτική και πλήρη απασχόληση. Αυτό είναι το καθήκον σας και ξέρω ότι θα το επιτύχετε και με τη δική μας την υποστήριξη επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των φιλελευθέρων ο κύριος Φερχόφστατ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Μάριο. Και εμείς της ομάδας Σπινέλη χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κατέχετε αυτή τη θέση. Είσαστε Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η εργασία σας, διότι σε λίγες εβδομάδες επαναφέρατε την Ιταλία στη σωστή οδό με πολλές μεταρρυθμίσεις απόλυτα αναγκές για τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη. Και έχουμε έναν μεγάλο φεντεραλιστή ενώπιόν μας εδώ από πλευράς Συμβουλίου. Δεν θα συνεχίσω στα Ιταλικά, μη φοβάστε. Ε, είμαι εξειδικευμένο στο Ιταλικό κρασί περισσότερο. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μάριο, ε, αυτό που χρειάζεται είναι κάτι περισσότερο από έπαινη σήμερα. Αυτό που χρειάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το ε, Συμβούλιο ασφαλώ είναι κάτι παραπάνω από ηθική υποστήριξη. Χρειάζεστε συγκεκριμένη υποστήριξη με ενδεχομένω ε, μια πρόταση μείωση των επιτοκίων για όλου στην Ευρώπη. Σήμερα, συνάδελφοι, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στην Ιταλία, ακόμα και μετά τις μεταρρυθμίσεις, ε, η Ιταλία πληρώνει τρεις φορές ε, παραπάνω επιτόκιο για τα δάνειά της από ότι η Γερμανία. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Οπότε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να συστήσουμε αυτό το Ταμείο Σωτηρίας, η γερμανική ιδέα, καλή ιδέα όμως, με 2,33 εκατομμύρια ευρώ και αυτό θα ήταν ένα ταμείο το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και για άλλων χωρών όπως της Γερμανίας. Και θα πρέπει να γνωρίζετε κύριε Μόντι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες σε ψηφισμά του κάλεσε να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Σωτηρίας του χρέους. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το ε, πακέτο των δύο μέτρων, το οποίο συζητούμε. Νομίζω ότι με αυτόν τον ε, τρόπο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις ε, τακτικές ενέσεις ε, χρημάτων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που είπατε για τα ε, ο, ομόλογα σταθερότητας. Χρειαζόμαστε όχι μόνο αλληλεγγύη, αλλά και ένα πραγματικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει ε, να ακολουθήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, τον κανόνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Χρειαζόμαστε μια πιο δομική λύση. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε κάνει. Ένα τρισεκατομμύριο ε, ευρώ έχουμε αφιερώσει για την επίλυση των κρίσεων. Τρεις χώρες είναι με πακέτα διάσωσης. Ε, έχουμε μείωση ε, της πιστοληπτικής ικανότητας τριών σημαντικών χωρών, Γαλλίας, Ιταλίας και ενδεχομένως Γερμανίας. Και παρόλα αυτά, δεν, βλέπετε, δεν, παρόλο το 1 τρισεκατομμύριο δεν έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Συνεπώς θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο εργαλείο για να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα των φορολογημένων. Ε, χρειάζεται μια διαθροτική μεταρρύθμιση της αγοράς ομολόγων στην Ευρώπη. Ε, τέλος, η Ιταλία δεν είναι η ίδια περίπτωση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ε, σήμερα θα πρέπει να δει τι κάνει η Ιταλία. Η Ελλάδα χρειάζεται διαφορετικέ αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται να μειώσει τον τεράστιο δημόσιο χρειάζεται να μεταρρυθμίσει το πολιτικό της σύστημα. Αυτά η Ελλάδα αφού τελειώσει τη δουλειά του στην Ιταλία ο κ. Μόντι, ίσως θα έπρεπε να σταλεί στην Ελλάδα. Θα ήταν ε, ίσως ένας εξαιρετικός μετακινούμενος πρωθυπουργός για όλες τις χώρες της, Ευρω... Ε, Ευρωζώνης που έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γκράτσιε, κύριε Φερχόφστατ. Και τώρα η κυρία Χάρμς, εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων. Γράτσια κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Μόντι, περνώ αμέσως στα γερμανικά. Με την ομιλία σας και όχι μόνο με το άρθρο που δημοσιεύσατε με τη συνάδελφο κυρία Σιλβί Γκουλάρση σήμερα, με την ομιλία σας νομίζω ότι διευκρινίσατε δύο πράγματα. Πρώτον, είστε εκείνος ο πολιτικός άνδρας που είναι σε θέση μετά από ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα να ε, εκπολιτήσει πάλι το κλίμα στην Ιταλία και μας δείξατε ότι θα μπορούσατε να είστε ένας από τους ισχυρούς πολιτικούς άνδρες που μπορείτε να εκπολιτήσετε ξανά και το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό γιατί περί αυτού πρόκειται. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την ομιλία σας και κάποιες, σε κάποια σημεία σκεπτόμουν ότι καλά είναι όλα αυτά, θα μπορούσαν όμως να είναι πιο ξεκάθαρα, πιο σαφή, ώστε να καταδειχθούν συγκεκριμένα οι δυσκολίες. Αναφέρθηκε η κατάσταση στην τελεία και από τον κύριο Φερχόφστατ, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία είναι χώρες όπου ο κόσμος φοβάται ακούγοντας τις ανταποκρίσεις από την Ελλάδα. Λέμε πάντα ότι η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα. Λέμε ότι η Πορτογαλία είναι διαφορετική, η Ισπανία είναι διαφορετική όπως και η Ιρλανδία. Αλλά γνωρίζετε ότι η κρίση δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο καθόλου, αλλά μπορεί να διαδοθεί και πριν από, λίγο, πριν από καιρό είδαμε ότι και στον τραπεζικό τομέα στις χρηματικές συναλλαγές η κρίση γιγαντώθηκε. Μπορούν λοιπόν να τεθούν κάποιες ερωτήσεις για να διευκρινιστούν από σας κάποια πράγματα. Πρώτον, κοιτάζοντας την Ελλάδα εσείς λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε πολιτική χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να διατηρήσουμε ενωμένη την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι με την πολιτική απέναντι στην κρίση όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί δεν είμαι βέβαιη ότι μπορώ, να απαντήσω καταφατικά. Η Νέλη Κρούσε, η Επίτροπος, είπε χθε ότι δεν θα ήταν και δράμα μεγάλο εάν ε, ε, ε, έβγαινε από την Ευρωζώνη η Ελλάδα πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η δήλωση αυτή. Τι θα πρέπει να σκεφτούν ε, πάνω σε αυτό οι Έλληνες μετά τη δήλωση αυτή. Μιλήσατε για πειθαρχία, δημοσιονομική πειθαρχία. Πιστεύετε εσείς ε, ως ένας πολιτικός που πρέπει να βάλει σε τα της Ιταλίας, πιστεύετε ότι είναι συνετή η δημοσιονομική πειθαρχία όταν στηρίζεται μόνο σε περικοπές, γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Ε, περικόπτουν, περιστέλουν και μόνο. Δεν νοικοκυρεύεται έτσι ένας προϋπολογισμός, ούτε έρχονται σε ισορροπία έσοδα και ε, δαπάνες. Παρά τις περικοπές βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας αυτής ε, βλέπουν επιδείνωση της κατάστασής τους. Οι φτωχοί ε, γίνονται φτωχότεροι. Πιστεύετε ότι είναι προοπτική εξόδου κρίσης αυτή που θα χρησιμεύσει και αλλού για άλλες χώρες. Και επειδή προέρχεστε από τον τραπεζικό τομέα, γιατί αποφασίσατε να πείτε ότι οι μεγάλες τράπεζες ε, είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν και πάντοτε θα πρέπει να αποδεικνύουν την ε, παρουσία τους και να καταξιώνονται παρόλες τις ε, αδυναμίες που, υπάρχει στο, υπάρχουν στο σύστημα αυτό. Νομίζω ότι προδιαγράφουμε ε, υπερβολικά αυστηρά την πολιτική των κρατών σε μικρότερη σημασία θέματα χωρίς, και παραγνωρίζοντας τα μεγάλα. Ενδεχομένως ε, ε, θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική προσέγγιση. Γνωρίζω ότι ε, αρχίσατε να λαμβάνετε μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. στην, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που δώσατε στην περίπτωση της Κορτίνα Δελπέτσο. Αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή συμφωνία που δεν θα επιτρέπει ε, αυτήν της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος περίπου 300 δις ευρώ ε, χάνονται με αυτόν τον τρόπο από τα έσοδα, φορολογικά έσοδα. Ε, διακόπτει ο ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υπομονή σας. Μία φράση μόνο θα μου επιτρέψετε στο τέλος, κύριε Μόντι. Μία, μία φράση μόνο. Κύριε Μόντι, εις ό,τι αφορά τους πρωθυπουργούς των χωρών της κρίσης βρίσκονται σε ιδιαίτερη κατάσταση γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, απολάβουν ιδιαίτερα μεγάλου σεβασμού και εσείς με την πείρα σας ε, ως ε, Επίτροπος έχετε ιδιαίτερη ε, ευθύνη σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης σε χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν αντιμετωπίσει κρίση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλαναν από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μην ξεχνάμε τους Monty Python, οι οποίοι μας ε, είπαν πάντοτε να βλέπουμε την λαμπρή όψη των πραγμάτων. Ε, αναφέρουν λοιπόν σε αυτούς τους άλλους Monty. Ε, τα οικονομικά νέα λοιπόν ε, είναι ζωφερά, πλην όμως ε, υπάρχουν ένας δυο λόγια να είμαστε αισιόδοξοι για την Ιταλία. Ε, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φερχόφστατ. Η Ιταλία ευτυχώς δεν είναι ίδια περίπτωση με την Ελλάδα. Όμως, η, η κακοδιαχείριση ήταν ένα φαινόμενο και της Ιταλίας. Ε, από πλεόνασμα Ιταλία σε 10 χρόνια πέρασε σε σημαντικό έλλειμμα. Και από ό,τι φαίνεται ότι προς το παρόν οι αγορές σέβονται τις ηγετικές σας Τα δεκαετή ομόλογα είναι μάλλον διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή χάρη στις ε, μεταρρυθμίσεις που έχετε προτείνει και κυρίως χάρη στη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, ε, που σας εξασφάλισε ένα χρονικό περιθώριο. Η, οικονομική, η δημοσιονομική εξυγίανση στην Ιταλία μπορεί να δουλέψει λοιπόν. Στην, στην Ελλάδα σίγουρα δεν δουλεύει. Ε, η η έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη θα ήταν ίσω κακή πολιτική για την Άγγελα Μέρκελ, αλλά νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη λύση για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Η δημοσιονομική εξυγένση θα διευκολύνει την κρίση, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για τι οικονομικέ μα αδυναμίε. Ε, ε, η, η απάντηση είναι η ανάπτυξη. Και έχουμε μια σειρά ε, εκκλήσεων πολιτικών ε, για υπέρ τη ανάπτυξης αλλά μέχρι τώρα έχουμε αποτύχει γιατί έχουμε εστιαστεί μόνο στα λόγια ε, και δεν έχουμε, δεν έχουμε κάνει τα λόγια πράξη. Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης είναι γραφειοκρατική και είναι η ίδια αντιμετώπιση που μας έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Βέβαια, υπάρχει ένα έγγραφο πολιτικής το οποίο εφαρμόζεται που είναι το έγγραφο του Μάριο Μόντι για την ε, ενιαία εσωτερική αγορά ε, το οποίο υποστήριξε τόσο πολύ ο κ. Χάρμπορ στην επιτροπή μα εδώ. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα τη Ευρώπη είναι ο ανταγωνισμός, ε, ο οποίο αντιμετωπίζεται δυστυχώ με εναρμόνιση και όχι με απελευθέρωση των αγορών. Η ενιαία αγορά έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πιο ευέλικτε αγορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση δεν είναι περισσότεροι κανόνες, περισσότερη ρύθμιση, περισσότερη γραφειοκρατία και εναρμόνιση και σίγουρα όχι περισσότερη Ευρώπη. Η απάντηση είναι μια καλύτερη Ευρώπη, μια Ευρώπη απελευθερωμένη ε, και ανταγωνιστική. Κύριε Μόντι, ω Πρωθυπουργό τη ε, Ιταλία, μιλώ για την ε, δημοκρατία. Βέβαια, εσεί δεν έχετε εκλεγεί από του πολίτε σα. Σίγουρα έχετε εκλεγεί από το Κοινοβούλιο τη Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πράξη αυτό το όραμα τη απελευθέρωση τη οικονομία και τη μεταρρύθμιση. Και όχι μόνο στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη. Αν πετύχετε σε, αυτή την, σε αυτό το δύσκολο έργο, θα έχετε του εξεπένους και την υποστήριξη όλων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάλλαναν Και τώρα εξ ονόματος ε, της ε, ε, ομάδας Γκουε της Αριστεράς ο κύριος Παδίκλη Γιαρίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβούμαι ότι για μία ακόμα φορά με τη συζήτηση αυτή προσπαθούμε να καλύψουμε, να καλουμουφλάρουμε ε, την ε, απίστευτη σκληρή θρησκεία που οδηγεί στην απώλεια την Ευρώπη, δηλαδή την λιτότητα. Δεν αναφερθήκατε στη λέξη αυτή κύριε Μόντι, αναφερθήκατε μονάχα στην πειθαρχία. Την είδαμε όμως την πειθαρχία και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η λιτότητα μπορεί να είναι θάνατος, ε, γιατί δεν επιτρέπει ούτε την οικονομική ανάπτυξη, ούτε την ανάπτυξη γενικότερα. Θυσιάζει την ευημερία των ανθρώπων ε, και το, κράτος, και το κοινωνικό κράτος μιλάμε για δικαιοσύνη. Τι είδους, δικαι... δημοκρατία, συγγνώμη, μιλάμε για δημοκρατία, τι είδους δημοκρατία, κύριε Μόντι για ποια δημοκρατία μιλάμε όταν ε, στην συμφωνία Europlus ε, μας ε, αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον διαπραγματεύσεις για τις συλλογικέ συμβάσεις. Ποια δημοκρατία όταν στις ερχόμενες συμβάσεις και συνθήκες βλέπουμε μονάχα ένα, μια διατύπωση που αναφέρεται μονάχα σε λιτότητα, σε πειθαρχία, σε μέτρα, σε περικοπές. Ποια δημοκρατία είναι αυτή. οι συνθήκες που γίνονται σήμερα δεν οδηγούν ούτε στην ανάπτυξη ούτε στην ε, ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Εμείς σαν ΓΚΟΕ κάνουμε προτάσεις και για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την απασχόληση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένα συζητήσει για τα θέματα αυτά. Εμείς θέλουμε προστασία της εργασία στην Ευρώπη. Θέλουμε το τέλος του κοινοβουλίου κοινωνικού και δημοσιονομικού και φορολογικού ντάμπινγκ. Θέλουμε πραγματική εργασία. Θέλουμε πραγματικές θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε πραγματικό φόρο ε, συναλλαγών στην Ευρώπη. Θέλουμε μια ουσιαστική πρόοδο και στο σύνορα όσον αφορά τις μεγάλες πρόοδους περιβαλλοντικές και άλλες. Θέλουμε να δώσουμε όθηση στην ε, βιομηχανία, στην έρευνα, στην ε, εκπαίδευση αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν εάν δημιουργηθεί ένα νέο οικολογικό και κοινωνικό ταμείο ε, το οποίο θα αντικαταστήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και που θα δώσει την ε, δυνατότητα να, βοηθήσουν, βοηθήσουμε πραγματικά τις ε, χώρες οι οποίες δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή γιατί θα είναι ένα ταμείο το οποίο θα δίνει 1% άμεσα στα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μην μου πείτε ότι υφιστάμενες συνθήκες σας δυσκολεύουν και δεν το επιτρέπουν, γιατί τις αλλάζετε τις υφιστάμενες συνθήκες κατά της βουλήσεως των λαών και κατά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. τον λόγο για την ομάδα τελευταία, ο κ. Σπερώνη. Κύριε Πρόεδρε Μόντι, εσείς βεβαίως ε, έχετε μεγάλες γνώσεις ε, για, περί τα οικονομικά ε, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη Λέσχη Μπίντελμπερκ και στα πανεπιστήμια, σε ακαδημαϊκούς κύκλους κλπ και πήγατε και στην ε, Wall Street ε, για να συναντήσετε αυτούς ε, τους χρηματοπιστωτικούς παράγοντες, αυτούς τους τραπεζίτες οι οποίες μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη Γιουρολάνδια. Αναρωτιέμαι, συναντηθήκατε με τους συνενόχους σας ή με τους κυρίους σας γιατί φαντάζομαι ότι και σαν παλαιός ε, επίτροπος συμφωνείτε με την ε, ε, οικονομική πολιτική που ακολουθείτε, άρα συνένοχος, ενδεχο... τους συνενόχους, άρα τους κυρίους σας ενδεχομένως, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προτίθεστε να καταλυστεύσετε τους φορολογούμενους, έτσι ώστε να βοηθήσετε και να στηρίξετε τους διεθνείς εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα η Ευρώπη δεν μας ανήκει, αν είναι έτσι όπως μας την ε, λέτε, ούτε τη θέλουμε. και δεν είναι δυνατόν όπως ε, ε, είπε και ο πρόεδρος Ναπολιτάνο να επιτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Μα θέλετε να βγείτε από την κρίση. Δεν είναι δυνατόν εσείς και οι ίδιοι με εσά, οι όμοιοι σας, δεν βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο φαλκιδεύετε την κατάσταση. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια Νορβηγία, μια Ελβετία, μια Νέα Ζηλανδία, ένας Καναδάς, μια Αυστραλία. Χώρες δυτικής δημοκρατικής παράδοσης. Χώρες των οποίων οι πολίτες χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς ευρώ βλέπουν την οικονομία τους και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε εμείς. Ευχαριστώ κύριε Σφερόνη. Okay. Okay. herr cohn bendit Κύριε Κονμένιτ, σα παρακαλώ. Το λόγο ο Γκόλνης. μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Βοντα, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, μάλλον το Συμβουλίου, όλοι χαιρετίζουν τη γρήγορη δράση σα και το σχέδιο λιτότητα ε, που μπορεί να ικανοποιήσει όλε τι απαιτήσει των συμπατριωτών ε, και πρώην, μάλλον του συμπατριώτη σα και πρώην διευθύνοντο τη ε, Goldman Sachs, του κυρίου Μάριο Ντράγκη, που τώρα είναι στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το έχουμε βέβαια το σχέδιο λιτότητα αναβαθμίσει σε σχέδιο διάσωση. Έτσι το έχουμε μετονομάσει. Πολύ θάρρο, πολύ στένο έχετε επιδείξει, αλλά τελικά, κύριε Πρόεδρο Συμβουλίου, υπάρχει συμβούλιο όταν από τη στιγμή που σε αυτή τη θέση γνωρίζετε ότι θα συνεχίσετε να ασκείτε αρμοδιότητε όπω και κατά το παρελθόν, χωρί ποτέ να σας ψηφίσουν ή να σας εκλέξουν, να υποστείτε δηλαδή ε, την εκλογική αναμέτρηση. Περιορισμένες λοιπόν ε, ε, οι εξουσίες που σας έχουν εκχωρέσει κάποιες σκοτεινές λέσχες όπως η λέσχη Bilderberg μπορεί να έχετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά δεν ξέρουμε τελικά τι νομιμοποίηση έχετε. Πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα. Όμως ε, όπως σας είπε ο κύριος Βόποντα που είναι Αυστριακός ή ο κύριος Φερχόφστατ ε, των Φιλελευθέρων ε, που είναι Φλαμανδός ε, σας απάντησαν αγγλικά σε αυτά που είπατε ενώ υπάρχουν διερμηνείς και δεν καταδέχθηκαν να χρησιμοποιήσουν την εθνική τους γλώσσα. Χρησιμοποίησαν τη γλώσσα του μεγάλου αδελφού, του Big Brother, των Βρετανών πατριωτών που κάθονται δίπλα μου.

σε εύθραυστη κατάσταση εισήλθε ε, σε αυτή την κρίση η Ιταλία και όταν αναλάβατε εσείς τα καθήκοντά σας. Από πρώτη μέρα όμως δείξατε την αποφασιστικότητά σας να, να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και ήδη έχετε εγκρίνει σημαντικά μέτρα. Αφενός το Δεκέμβριο στην Ιταλία πέρασε ένα νέο ε, πακέτο λιτότητας ε, για την εξηγήνωση των οικονομικών της Ιταλίας που θα επιτρέψει στη χώρα να επιτύχει ήδη από το 2013 ένα πολύ σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και να μειώσει το χρέος της χώρας. Επίσης ε, το τελευταίο καλοκαίρι αλλά και μέχρι τις προηγούμενες εβδομάδες ε, λήφθησαν πολλά μέτρα για τις συντάξεις, ε, τη φορολογία, τον ανταγωνισμό, το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Τα πιο πρόσφατα μέτρα για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων ε, και τη διοικητική απλούστευση σίγουρα θα συμβάλλουν και αυτά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έροντας φραγμούς προς το εμπόριο και μεγαλώνοντας την δυνατότητα προσαρμογής της χώρας η Κομισιόν, για να ολοκληρώσω, χαιρετίζει τι αποφασιστικέ δράσει και ενέργειε ε, τη Ιταλική κυβέρνηση και στέκεται στο πλευρό τη για να την στηρίξει, να την βοηθήσει ε, όταν και ε, με όποιο τρόπο το κρίνει απαραίτητο η Ιταλική κυβέρνηση. Ένα σαφέ παράδειγμα είναι η βοήθεια τη Κομισιόν για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων με την δημιουργία μια ομάδα ειδική που θα βοηθήσει την Ιταλία και για τη χρήση των δραστηριοτήτων μέχρι το 2013. Όπω ε, θα είδατε ίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε την ε, ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι έχετε πολλού ε, φίλου, θα έλεγα και οπαδού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εύχεται στην Ιταλία, στην κυβέρνησή σα, αλλά και σε, εσά προσωπικά, κάθε επιτυχία στι προσπάθειέ σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφκοβίτσου. Θα να δώσω λόγο στον ε, Πρωθυπουργό κ. Μόντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια και μίλησα περισσότερο στην πρώτη μου παρέμβαση και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος στα δύο συμπερισματικά λόγια τα οποία θα πω ξαναευχαριστώντας σε εσά κύριε Πρόεδρε καθώς επίσης και τους βουλευτές που θέλησαν να εκφράσουν την στήριξή τους ε, καθώς επίσης και την εκτίμησή τους για τη χώρα μου και για μένα προσωπικά. Αυτά τα λόγια, η έκφραση των συναισθημάτων αυτών και οι πράξεις τους μας ανακουφίζουν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε την Ιταλία ε, για να μπει σε μια πραγματική αναπτυξιακή και ευρωπαϊκή τροχιά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς για τα σχόλια τα οποία έκανε. Θα απαντήσω μονάχα σε δύο σημεία και επιφυλάσσομαι να μελετήσω στο γραπτό μεταφρασμένο κείμενο λόγω των υπαρξιακών φιλοσοφικών στοιχείων που ανέφερε ε, ο κύριος Σπερώνη, για, τον οποίον όμως, για τα οποία όμως λόγια του τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Σύντομα λοιπόν, σύντομη απάντηση, μάλλον ε, σε αυτήν την παρατήρηση του κυρίου Γκόλνης, στον οποίο θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να καυχηθώ Ε, δεν μπορώ να καυχηθώ λοιπόν ότι έχω ε, αυτήν την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση που έχουν οι άμεσα εκλεγμένοι όπως εσείς. Βεβαίως εγώ ποτέ δεν υπέβαλα τον εαυτό μου σε αυτήν την διαδικασία. Μου πρότειναν μία θέση την οποία δεν θα έπαιρνα από μόνος μου και αυθορμήτως. Εάν σας ζητούσα να παρέμβετε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση ε, ως επικεφαλής ε, της κυβερνήσεως στη χώρα σας ε, θα είχατε αρνηθεί λέγοντας ότι θα το κάνατε μονάχα εάν είχατε δημοκρατική νομιμοποίηση. Φαντάζομαι ότι μόνο αυτό θα κάνατε εσείς κύριε Γκόλνης. παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου, οι διερμηνείς δεν τους ακούν δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ και ε, για αυτό τον έντονο τρόπο και τα συναισθήματα τα έντονα με τα οποία με υποδεχτήκατε. Ε, κύριε Χάρμσον ξεκινώντας, ε, παίρνοντας μάλλον σαν έναυσμα την, την ε, παρέμβασή σας. Έγιναν πάρα πολλά σημαντικά σχόλια σε σχέση με την ε, ελληνική κρίση. Όλοι σκεφτήκαμε πάρα πολύ όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας. Εγώ, μια και είμαι από τους πρεσβύτερους μεταξύ ημών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δούμε ιστορικά τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως, η ομότητα, η σκληρότητα με την οποία να αντιμετωπίζεται τούτη τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να μας οδηγήσει στο να θεωρήσουμε την παρέμβαση αυτή υπερβολική και ενδεχομένως να είναι. Όμως, να μην λησμονούμε ότι για πολλά χρόνια η ελληνική πολιτική, και το λέω σαν απλός εξωτερικός παρατηρητής και με μεγάλη μετριοφροσύνη, αποτέλεσε τον ε, καλύτερο, τον τέλειο κατάλογο των κακών πρακτικών. και το άρθρο αυτό αναφέρεται και στο άρθρο που ανέφερα και εγώ προηγουμένως όταν λέμε ότι στην Ευρώπη λειτουργεί η δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο αλλά δυστυχώ όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ουσία ε, εδώ διαψεύδεται αυτή η αρχή εδώ έχουμε ευρωπαϊκό επίπεδο δημοκρατίας από την άλλη πλευρά ε, δεν θέλω να ε, θεωρήσουμε σαν υποδείγματα καλή δημοκρατία αυτά τα οποία είδαμε στην Ελλάδα ή σε άλλε χώρε. δηλαδή οπωσδήποτε βασιζόμαστε σε ε, πελατειακή δημοκρατία, σε πελατειακές διαδικασίες, σε νεποτισμό, ε, σε διαφθορά διευρυμένη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, έστω και αν κρίνομαι ως ε, υπερβολικές ε, τις λιτότητες γενικά τις οποίες επιφέρει ε, η ευρωπαϊκή παρέμβαση, θα ήθελα και, και εγώ μάλιστα εν παρόδο να σας πω ότι κάποια στιγμή θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή η λιτότητα. Αυτή η παράδοση διαρκούς λιτότητας της Γερμανίας, την οποία λίγο όλοι μας αφορούν, αφομοιώσαμε μέσω του ευρώ μπορεί να βοηθήσει ε, την ε, πολιτική κάποιων χωρών. Γιατί ξέρετε στο παρελθόν ήταν ίσως λίγο πολύ εύκολο στους πολιτικούς να λένε ναι σε οποιαδήποτε απέτηση, οποιασδήποτε συνδεχνίας ε, υπονομεύοντας το μέλλον των μελλοντικών γενεών, υπονομεύοντας την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα τους. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι ενδεχομένως φτάσαμε πλέον στο άλλο άκρο, στο ίστατο άκρο της ε, λιτότητας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον αυτό το εκρεμές άρχισε να κινείται μετακινήθηκε από το άλλο άκρο στο οποίο βρισκόταν, ακόμα και στη χώρα μου βεβαίω. Και ελπίζω ότι θα έχει βοηθήσει κατά αυτή την έννοια η μεγαλύτερη πειθαρχία. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ για όσα μας είπατε. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση.